ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι προς την Γιούλια Τιμοσέκο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στη δήλωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν σε σχέση με το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας. Θα ήθελα να καλωσορίσω με μεγάλη χαρά ως πρώην συνάδελφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την κυρία Τόνικ Σμιτ. Έχετε το λόγο. Ε, καλώς ήρθατε κυρία Πρωθυπουργέ. Σας δίνω λοιπόν το λόγο ε, για, το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας. Έχετε το λόγο, κυρία Τόνικ Σμιτ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε,